Καλησπέρα σας, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Έχουμε ένα δύσκολο θέμα να συζητήσουμε την ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Ελεκτρονικών Επικοινωνιών. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Πέτρα Κάμερεβέρτ και έχει συντάξει μια έκθεση για τις σχέσεις μεταξύ των υπήρων Το θέμα είναι πολύ δύσκολο. Για, μη, ε, για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πολύ καλά αυτά τα θέματα, ίσως να είναι και λίγο δύσκολο να κατανοήσουν την πέτρα. Πάντως, ε, με τον τρόπο αυτό κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα προς την αγορά των ε, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των υπηρεσιών των σχετικών, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην ανοίξουμε διάβλατα τις πόρτες σε κάτι που πάντοτε θέλαμε να αποφύγουμε. Ουδετερότητα, κατανομή συχνοτήτων, προστασία προσωπικών δεδομένων, αυτά πρέπει να τα διατηρήσουμε. Στόχος μας είναι να είμαστε με την Επιτροπή ΙΜΚΟ ισότιμες επιτροπές 50-50 και τελικά επειδή υπάρχει τρίτη επιτροπή θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο στενά συνδεμένες εργασίες, άρα είναι 49-9 κατά κάποιο τρόπο η εκπροσώπηση. Äh, Θα προσέξουμε πολύ να μην ε, πέσουν στον κάθο να χρήσουν οι προτάσεις που θα διατυπώσουμε. Αν δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα στη συναπόφαση, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πρόταση που ελπίζουμε να μπέσει, όπως είπα, στον να χρήσουν. Πέτρα, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Ντόρις, αγαπητοί συνάδελφοι. όταν γίνεται λόγος για το ψηφιακό θεματολόγιο, πιο πολύ πρόκειται για το τεχνικά εφικτό. Δηλαδή, τι ταχύτητε για το διαδίκτυο μπορούμε να εξασφαλίσουμε, αλλά δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πιο σημαντικά ζητήματα από τα αμυγό τεχνικά. Υπάρχουν θέματα οικονομικής ανάπτυξης, ανεργίας και σήμερα μιλάμε για την δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ε, τηλεπικοινωνιών. Πάλι όμως ε, για περισσότερα πρόκειται και δεν είναι μόνο θέματα αγωνιστικότητας. Ποια είναι η δική προσωπική άποψη. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σταυροδρόμι στην ψηφιακή αυτή επανάσταση. Θέλουμε ε, έναν ψηφιακό κόσμο που θα είναι πώς ακριβώς. Θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Ή να πιστεύουμε ότι έχουμε τελικά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Θέλουμε να ζούμε σε έναν κόσμο που καταγράφονται τα πάντα, που ελέγχεται ε, ε, και καταγράφεται το κάθε βήμα που κάνει ο καθένας από εμάς. Μιλάμε για ελευθερία επικοινωνιών, μιλάμε για πρόσβαση, μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα και για τη συμμετοχή στην κοινωνία μας σε τελική ανάλυση. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα και στους συμπολίτε να συμμετέχουν σε αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες. Πιστεύω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε την πρόσβαση των πολιτών στο διαδικτύο από πλευράς περιεχομένου, και ουδετερότητας δικτύου. Είναι κάπως τεχνοκρατικός ίσως αυτός ο κανονισμός, αυτή η ρύθμιση, έτσι θα σας ακούγεται φαντάζομαι, αλλά πίσω από τον τεχνοκρατικό τίτλο υπάρχουν κομβικά σημεία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κατά την άποψή μου πρέπει να βρούμε απαντήσεις ώστε να οδεύσουμε προς μία κατεύθυνση με ελευθερία επικοινωνίας, με ελευθερία επιλογή και ακόμη και αν η πρότασή μας δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένη προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύουμε. Να σας πω κάποια σημαντικά στοιχεία. Στην Επιτροπή Πολιτισμού ε, το θέμα της περιαγωγής, ε, του να μην υπάρχει περιαγωγή, ε, είναι θέμα που δεν μας αφορά ακριβώ. Δεν καταθέσαμε λοιπόν τροπολογίες γιατί είναι αρμοδιότητα πιο πολύ άλλων επιτροπών. Άρα επαναλαμβάνω καμία τροπολογία από πλευρά μας. Έπειτα έχουμε την πολιτική των συχνοτήτων, την πολιτική του φάσματος. Νομίζω ότι πέρυσι ασχοληθήκαμε διαμακρών με το θέμα αυτό. Θέλαμε να περάσει και η άποψη της Επιτροπής Πολιτισμού στο Κοινοβούλιο. Τελευταίο θέμα είναι η ουδετερότητα των δικτύων. Εκεί ε, και στο δεύτερο έχω επικεντρωθεί πιο πολύ, γιατί πιστεύω ότι αυτά είναι και τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εμάς. Επηρεάζουν την ελευθερία επιλογής και επικοινωνίας. Αυτά είναι για μας τα πλέον ενδιαφέροντα. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό, αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν γίνει νόμος θα επηρεάσει τον πλουραλισμό, την πολυμορφία την πολιτισμική, την πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης, την ενημέρωση. Και σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του τελευταίου πακέτου επικοινωνία στα κράτη-μέλη, γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή του τελευταίου πακέτου τηλεπικοινωνιών, τουλάχιστον 100%. Η Κομισιόν Επίσης φαίνεται να παραγνωρίζει και τα απορίσματα της δικής της ε, Επιτροπής Εμπειρογνωμών. Σύγκληση του κακουστικού κόσμου. Ε, μόλις άρχισαν να το αξιολογούν το θέμα. Το συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Απαντήθηκαν τα ερωτήματα, δεν τα έχει αξιολογήσει όμως ε, τα απορίσματα η Κομισιόν. Και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το δούμε και στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου κανονισμού. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη επαρκών κινήτρων για επενδύσεις στο δίκτυο. Και αν δεν επιληθεί αυτό το πρόβλημα, δεν έχει και νόημα να ασχοληθούμε μετά του φάσματος. Γιατί θα προκύψουν προβλήματα που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσβαση και το περιεχόμενο. Επομένως, Η ελευθερία επικοινωνία και ενημέρωση επίσης θα πληγεί, θα επηρεαστεί. Ουσιαστικά επαναλαμβάνω τα όσα περιλαμβάνει η θέση μας ε, για τις ραδιοσυχνότητες. Είπαμε ότι οι ραδιοσυχνότητες είναι ένα δημόσιο αγαθό. Άκρο σημαντικό λοιπόν για την εκπλήρωση σημαντικών κοινωνικών καθηκόντων. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το θέμα αυτό στην όλη συζήτηση για τις ραδιοσυχνότητες. Πρέπει να αποτελέσει τη βάση της πολιτικής της Ένωσης για τις ραδιοσυχνότητες. Τώρα, κατά πόσο ο κανονισμός είναι σωστή νομική βάση, δεν νομίζω, δεν συμφωνώ. Υπάρχουν επίσης διαφορετικά ζητήματα περιφερειακά, τοπικά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και κατά την άποψή μου τα κρατημέλη θα πρέπει να έχουν και αυτά την δυνατότητα να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούν τις ραδιοσυχνότητες και για κοινωνικά και για πολιτισμικά καθήκοντα. Ο φορέας ο οπτικοακουστικό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί για δημιουργική οικονομία, για θέατρο, για διάφορους στόχους αυτές τις συγνώτες. Και αν αυτά τα αισθήματα δεν τα λάβουν υπόψη μας θα δημιουργηθούν προβλήματα. Αυτά όλα λοιπόν προσπάθησα να τα καλύψω με τις ε, τροπολογίες μου 2 και 3. Και πολύ σημαντικό είναι το δικαίωμα των κρατών μελών να υλοποιεί μέτρα ώστε οι ραδιοσυχνότητες να μπορούν να χρησιμοποιούνται για πολιτισμικούς, ε, πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η Κομισιόν τώρα, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να έχει το ρόλο του συντονιστή, του αρρωγού, όταν υπάρχει πρόβλημα, μια αντιπαράθεση ή σύγκρουση μεταξύ των μελών. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε 700 ζώνες συγνωτήτων Πρέπει να δούμε τι ακριβώ θέλει να κάνει η Κομισιόν. Θέλει να απαγορεύει, θέλει να ελέγχει τα μέτρα που θα προτείνουν ή θα υλοποιούν τα κράτη-μέλη. Οι συχνότητα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Χρήστε των ραδιοσυχνοτήτων. Στο δίκτυο πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πρέπει να αναπτύξουμε νέων εξοπλισμό, Πιο εύρωστο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει βέλτιστη χρήση των δύο συχνοτήτων προς όφελος όλων των πλευρών. Hier kann man wirklich auf der Selbstregulierung Ίσως η αυτορύθμιση θα ήταν πιο καλή προσέγγιση. Ίσως θα έπρεπε να διαβολευτούμε με τους ε, εμπλεκομένους φορείς, αλλά αυτό δεν το βλέπουμε ως πρόταση. Ένα δεύτερο τμήμα λοιπόν των δικών μου προτάσεων είναι πώς θα εξασφαλίσουμε την ευθερότητα του δικτύου. Όλοι μας συμφωνούμε ότι το διαδίκτυο έχει τεράστιο δυναμικό για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το μέσο αυτό να παραμένει ανοιχτό ελεύθερο. Να έχει βέβαια μια εύρωστη αρχιτεκτονική και δομή που δεν θα επιτρέπει διακρίσεις από κανένα και προς κανένα συμμετέχοντα ή περιεχόμενο και θα μπορούν όλοι να συμμετέχουν ενεργά. Ουδετερότητα δικτύου λοιπόν. Θεμελιώδης για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό, το τεράστιο αυτό δυναμικό του διαδικτύου πρέπει να είναι ανοιχτό και να μην οδηγεί σε διακρίσεις. Είναι ένας μοχλός καινοτομία για τις κοινωνίες μας για οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Ουδετερότητα λοιπόν δικτύου για την πολυμορφία, τον πλουραλισμό. Πρέπει να υπάρχει συνιστόσα ισότιμων ίσων ευκαιριών. Να προστατεύονται οι ίσες ευκαιρίες. Γιατί αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε για την ελευθερία έκφρασης και για την πολιτισμική και πολιτιστική πολυμορφία. Είναι ένα δημόσιο αγαθό το διαδίκτυο. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην το αφήσουμε στο έλο ε, των αγορών και των δυνάμεων των αγορών. Αν θέλουμε λοιπόν ε, να έχουμε ένα ανοιχτό ελεύθερο διαδίκτυο προσανατολισμένο στην καινοτομία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από διακρίσεις. Λόγω εφαρμογών περιεχομένου δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο στο περιεχόμενο του διαχειριστέ. Εκεί έγκυται λοιπόν η ιδιαιτερότητα. Και αυτά προτείνουμε στην έκθεση. Δεν θέλουμε να έχουμε κατάρριξη της ιδιαιτερότητας και να διαδίκτυο διπλών δύο ταχυτήτων. Επίσης η Κομισιόν κάνει πολλές προτάσεις για τις ειδικέ υπηρεσίες που όμως ναι, να υπάρχουν αλλά παράλληλα προς το διαδίκτυο. Πρέπει να είναι ξεχωριστές. Δεν πρέπει να περιορίζουν ε, τον ανοιχτό χαρακτήρα του διαδικτύου. Και θα πρέπει η πρόσβαση στο διαδίκτυο να γίνεται σύμφωνα με την αιχμή της τεχνολογίας. Διαχειριζόμενες υπηρεσίες, ναι, να υπάρχουν managed services, αλλά όχι σε βάρος των χρηστών και του ανοιχτού δικτύου που θέλουμε. Και θα πρέπει να επακολουθείτε εκ του σύνεγγυς ε, πολύ αυστηρά η δημιουργία αυτών των ε, δικτύων. Την ουδετερότητα την έχουμε ήδη συζητήσει Έχουμε συζητήσει και τα περιπαιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Πρέπει να βρούμε έναν καλό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με την πρόταση όπως αυτή περιλαμβάνεται στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής. Έχω δει το άρθρο 19 και 23 πολύ προσεκτικά. Εκεί γίνεται λόγος για διακρίσεις ε, περιεχομένου, γίνεται ράση προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τα μεταδεδόμενα δεδομένα. Αυτά ουσιαστικά στρέφονται κατά της ιδιαιτερότητας του δικτύου. Ανησυχούμε με αυτές τις προτάσεις. Φοβούμαστε ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την ελευθερία των ε, μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία έκφρασης. Στις τροπολογίες μου λοιπόν έχω προσπαθήσει ξεκάθαρα να τοποθετηθώ πάνω σε συγκεκριμένα σημεία. Μη διακριτική μεταχείριση των πακέτων δεδομένων, ανεξαρτήτως προέλευσης προορισμού περιεχομένου και γενική υποχρέωση διαβίωσης των πακέτων δεδομένων σε ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας από όλους τους χειριστές του διαδικτύου που θα πρέπει να τηρούν την αρχή της ε, βέλτιστης προσπάθειας. Να μην είναι σε βάρος ε, της ποιότητας η ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται ή δεν θα πρέπει να επιτρέπεται έλεγχος των πακέτων, επιθέωση των πακέτων. Η διαχείριση θα πρέπει μόνο για τεχνικούς λόγους να επιτρέπεται. Οι ειδικέ υπηρεσίες, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε κλειστά συστήματα και δίκτυα. Τελείως δηλαδή έξω από το διαδίκτυο. Ξεχωριστά από το διαδίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να περαστούν περισσότερα καλώδια αν θέλετε. Απλά θα υπάρχουν διαφορετικά πρωτόκολλα χειρισμού. Δεν θα γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου του διαδικτύου ο έλεγχος αυτών. Θέλουμε να είναι ανοιχτό το διαδίκτυο. Και αν οι χειριστέ πολλούν τέτοιου υπηρεσίε υπηρεσίες, θα πρέπει ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν υποχρέωση να παρέχουν και μία ε, υπηρεσία ανοιχτή πρόσβαση. Οι χειριστές δηλαδή πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να παρέχουν μόνο αυτές τις εξειδικευμένες υπηρεσίες γιατί τότε θα συρρυκνωθεί το ελεύθερο διαδίκτυο. Το βλέπουμε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, το βλέπουμε να συμβαίνει ήδη σε κάποιες χώρες εκεί. Εκεί βλέπουμε τι μορφή μπορούν να πάρουν αυτές οι εξειδικευμένες υπηρεσίες. Σε μια πύλη ή στο Google κάποιες προσφορές συγκεκριμένε, εφημερίδες, αν υπάρχουν εξειδικευμένε υπηρεσίες, ε, αυτές οι μαζικές πληροφορίε που μπορεί μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες. Δεν θα πρέπει να παρακαμφθεί το διαδίκτυο γιατί ε, αυτό θα είναι πραγματικά κρίμα. Θα βλάψει την καινοτομία θα μειώσει τις οικονομικές ευκαιρίες και δυνατότητες που έχει το διαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά τη νομική μορφή, δεν νομίζω ότι ο κανονισμός ε, είναι ιδέως νομική μορφή. Υπάρχει έλλειψη σαφήνειας. Σε πολλά κομμάτια του κειμένου ε, πραγματικά δεν καταλαβαίνει κανείς που το πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ισχύει ιδίως για το άρθρο 19. Στην αρχή νόμιζα ότι εγώ κάποιο πρόβλημα έχω και δεν καταλαβαίνω. Αλλά μετά απευθύνθηκα σε πολλού ενδιαφερομένου φορεί από διάφορα υπόβαθρα και του ζήτησα να μου εξηγήσουν τι λέει τελικά αυτή η παράγραφο, τι σημαίνει. Και τελικά οι περισσότεροι, ενώ όχι όλοι, μου είπαν ούτε εμεί καταλαβαίνουμε τι προτείνει η Κομισιόν. Άρα θα πρότεινα το αν άρθρο και οι λόγοι οι σχετικοί με την ύπαρξή του να απαλληφθούν, να διαγραφούν. Διότι δεν νομίζω ότι είμαι στους βουλευτές θα πρέπει να καθίσουμε να προβαίνουμε σε ερμηνείες για το τι ενδεχομένως εννοούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν είναι σαφές, αν δεν είναι σαφής ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε, δεν έχουμε παρά να διαγράψουμε αυτή την παράγραφο. Και αν η Κομισιόν το επιθυμεί, σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις μπορεί να μα εξηγήσει σαφέστερα τι εννοεί. Και εμείς να συμφωνήσουμε ή να μην συμφωνήσουμε, και αν συμφωνήσουμε να το βάλουμε ξανά στο κείμενο δεν, βοηθάει την, ε, σάφια, την, ε, την ε, νομική σαφήνεια όταν δεν καταλαβαίνει κανείς περί τίνος πρόκειται. Θα ήταν ευπρόσδεκτο φυσικά η Κομισιόν να αποσύρει την πρόταση αυτή. Και στο πλαίσιο της κανονικής διαβούλευσης να συζητήσουμε όπως πρέπει το όλο θέμα και με βάση αυτό να συντάξουμε ή να συνταχθεί τέλο πάντων μια νέα ισορροπημένη πρόταση για την αγορά τηλεπικοινωνιών. Αν λοιπόν είναι σημαντική η περιαγωγή, διαγράψτε αυτό το κείμενο, κάντε μια πρόταση συγκεκριμένη, κομισιόν, Μήπως θα ήταν καλό και λίγο πριν τις ευρωεκλογές θα ήταν καλό για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, να το συζητήσουμε. Αν τώρα η Κομισιόν όμω αρνηθεί και πει ότι είναι πακέτο και ω τέτοιο μόνο μπορεί να ισχύει, δεν μπορούμε να βγάλουμε μόνο δηλαδή τα τη περιαγωγή. Τι γίνεται άμα βγει η περιαγωγή. Νομίζω ότι τη στάση τη Κομισιόν δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε σε ό,τι αφορά αυτά που θέλει να κάνει για την περιαγωγή. Παρότι δεν είναι το δικό μα θέμα ω Επιτροπή. Τίθεται και το θέμα των συχνοτήτων. Σα τα είπα και πριν. Πρέπει να τα διατυπώσουμε πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Να μην καταστρέψουμε με τα χέρια μα αυτά που πασχίσαμε να δημιουργήσουμε τόσο καιρό. Ουδετερότητα δικτύου. Οι προτάσει δεν θα οδηγήσουν σε ουδετερότητα δικτύου, αλλά εμείς θέλουμε να προωθήσουμε έναν οργανισμό που θα στηρίζει την ουδετερότητα του δικτύου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρα. Ήταν όλα ξεκάθαρα. Ε, σε αυτά τα τρία σημεία να περιοριστούμε, τα έχεις ε, περιγράψει με μεγάλη σαφήνεια στο έγγραφό σου, στο κείμενό σου. Και εγώ βλέπω τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, όπως και εσύ. Η κυρία Φέρχαϊμ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ξεκάθαρη εισαγωγή, για τον ξεκάθαρο και σαφή τρόπο που παρουσιάσατε τις ε, θέσεις σας και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είχαμε μια καλή διαδικασία συναπόφασης, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον πολιτισμό. Νομίζω ότι ως Επιτροπή πρέπει να δώσουμε προσοχή στα δικαιώματα που ενέχονται. Ε, όχι να, δίνουμε, να δώσουμε απλώς τη γνώμη μας. Πρέπει να υπάρξει τριμερής διάλογος, πρέπει να συνεργαστούμε με τις συναρμόδιες επιτροπές, να ισότιμα να συμβάλλουμε στη λήψη της απόφασης και ελπίζω ότι η δική μας άποψη θα προαχθεί. Ε, ξαφνιάστηκα κιόλα σήμερα το πρωί στη συζήτηση, χωρίς μια κατάλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων, χωρίς μια σωστή διαδικασία διαβούλευση έχουν γίνει όλα αυτά. Δηλαδή μας παρουσιάζονται κάποια στοιχεία έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο αντίκτυπος στον τομέα του πολιτισμού είναι τεράστιος για την περιαγωγή θα ήταν πάρα πολύ καλό να μπορέσουμε να δείξουμε στους πολίτες πριν από τις νέες ευρωεκλογέ ότι βοηθούμε και αλλά μπορούμε να, να, θυσιάσουμε το θέμα της περιαγωγής εάν θεωρούμε πως δεν έχει προσεγγιστεί με το σωστό τρόπο. Για την ουδετερότητα του δικτύου, για την ανοιχτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι θέματα πολύ σημαντικά, αλλά λείπει η σαφήνεια για το κατά πόσο, για τον βαθμό στον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι εξειδικευμένες υπηρεσίες ε, ανώτερου επίπεδου. Ε, σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμε στον ιατρικό τομέα, για παράδειγμα. Εκεί που τα νοσοκομεία θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ε, χρειάζονται πραγματικά ένα δίκτυο με ποιότητα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στο μέσον μιας εγχείρησης, επειδή καταραίει το διαδίκτυο. Αυτό είναι αλήθεια και το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που να είναι ανεξάρτητο από το ελεύθερο και προσβάσιμο διαδίκτυο. Θα πρέπει να βασίζεται στις δυνατότητες μετάδοσης και αναμετάδοσης. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και ένα υλικό ε, δίκτυο δεν είναι δυνατόν να περιορίζουμε το ανοιχτό διαδίκτυο για να επιτύχουμε αυτό. Δεν θέλουμε να υπερκεράσουμε, να παραγωνίσουμε το ελεύθερο και ανοιχτό ε, διαδίκτυο. Θα πρέπει αυτό να περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό τμήμα ε, του φάσματος. Ε, εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία, να δώσουμε μεγάλη σημασία στο πώς θα χειριστούμε το εύρος των συχνοτήτων. Πολλές φορές στις αγροτικές περιοχές έχεις μόνο ένα διακομιστή και έχεις μόνο μία δυνατότητα. Ε, πο, πολλές φορές υπάρχει μια δέσμη υπηρεσιών, το καθεαυτό ίντερνετ και οι άλλε μαζί, οπότε δεν υπάρχει και ανταγωνισμός βασικά θέλουμε να έχουμε μία αγορά με ανταγωνισμό. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχουμε αρκετές δικτυακές υποδομές και δεν έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό σε πάρα πολλούς ε, τομείς και αυτό ισχύει και για τους παρόχους περιεχομένου, για τα μέσα, για τον κόσμο του θεάματος, για τον κόσμο των δημιουργών. Υπάρχουν αυτές οι εξειδικευμένε υπηρεσίε, αν υπάρξουν αυτέ οι εξειδικευμένε περιουσίε, υπάρχει ο κίνδυνο να μην είναι διαθέσιμε τελικά στο κοινό. Ε, το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο μέσω του ελεύθερου και δωρεάν διαδικτύου, όπως γίνεται μέχρι τώρα και θα πρέπει να διατίθεται και στη σωστή ποιότητα. Αν έχουμε μια εξειδικευμένη υπηρεσία και μια υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία και έχεις μια ειδική σύμβαση με την υπηρεσία τηλεπικοινωνιών, τότε θα πρέπει είτε να, οι υπηρεσίες να παρέχονται μέσω του διαδικτύου ε, σε συμβατική βάση ε, και το, η σχετική σύμβαση θα πρέπει να ορίζει τους όρους ποιότητας. Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στον πολιτισμό γιατί πρέπει να δούμε και πώς θα συντάσσονται οι σχετικές συμβάσεις. Οπόμενος πρέπει να, θα πρέπει να υπάρχει για παράδειγμα μια ελάχιστη ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων, μια, ένα ελάχιστο εχέγγυο ποιότητας των δεδομένων. Τα, οι σχετικές συμβάσεις θα πρέπει να, να αιτιολογούν το ανώτατο όριο της ε, ποσότητας ή της ταχύτητας μετάδοσης διαβίβασης των δεδομένων. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε έναν συνδυασμό εξειδικευμένων ή διαχειριζόμενων υπηρεσιών ή ελεγχόμενων υπηρεσιών και του ελεύθερου και ανοιχτού διαδικτύου. Έτσι ώστε στο μέλλον ε, οι συμβάσει που θα συνάπτουν οι συνδρομητέ με του ε, διακομιστέ ή με του φορεί, ε, με, τους, με τι επιχειρήσει, θα πρέπει να θεσπίζουν με σαφήνεια τα σχετικά με τα στοιχεία. Δηλαδή θέλω να ξέρω πόσα δεδομένα και πόσο χώρο έχω μέσω των εξειδικευμένων, των εξειδικευμένων υπηρεσιών ή τι χώρο και τι δυνατότητες έχω μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών, ε, συχνότητες. Υπήρξε ένα κείμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, ένα έγγραφο, που λέει ότι μέχρι το 2015 θα πρέπει να έχουμε ένα εύρος ζώνης ε, να έχουμε επιτύχει μια ευρυζωνικότητα μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Θα πρέπει βεβαίως να δοθεί χώρος στις τηλεπικοινωνίες και θα πρέπει να γίνει και μια σωστή κατανομή. Σύμφωνα με κριτήρια ποιότητας και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα δοθεί τελικά περισσότερο στο, στις ραδιοσυχνότητες ή στην κινητή τηλεφωνία. Πρέπει όμως ότι αυτό το, τα 800 οι 800 συχνότητες που έχουμε να διατεθούν και να κατανεμηθούν με σωστό τρόπο, έτσι ώστε και οι τηλεπικοινωνίες να έχουν αυτό που τους χρειάζεται. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Σε κάποιους τομείς μάλλον εάν τα κράτη-μέλη ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, θα ε, πάνε όλα καλύτερα. Αν απελευθερωθούν ε, οι 700 ραδιοσυχνότητες για τη ραδιοτηλεοπτική ε, μετάδοση, θα πρέπει να δούμε πώς τα κράτη-μέλη θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Το Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε, δεν πρέπει να ξεχνά τι έχει γίνει στο παρελθόν και να παρακολουθεί την κατάσταση στην περιαγωγή, όσο αφορά την περιαγωγή. Πριν από ένα χρόνο είχαμε την περιαγωγή 3 ε, για τις επιχειρήσεις, ε, για τον ανταγωνισμό. Είχαμε λοιπόν ε, χωριστές συμβάσεις για την περιαγωγή με καινούργιες τεχνολογίες. Και αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τα μέσα του 2050. Το 2015, με συγχωρείτε. Ε, και τώρα κάποιοι μιλούν για το 2016, γιατί δεν είναι δυνατόν να μετακυλιστεί και όλο το κόστος στους τελικούς χρήστες. Ε, αν δει κανείς τα τιμολόγια σε κάθε χώρα, θα δει ότι δεν, είναι, δεν υπάρχει διαφάνεια. Ε, το, το κόστος ε, της περιαγωγής ε, για έναν πάροχο δικτύου, για έναν διακομιστή, είναι κάτι που κρατείται μυστικό στην εταιρεία και δεν υπάρχει διαφάνεια. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό θέμα για μας σήμερα, ήθελα απλώς να το θίξω. Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο έγγραφο πρέπει να δούμε πώς θα, τι θα πούν οι άλλες επιτροπές, η Επιτροπή Ήτρα, τι θέλει να αφαιρέσει, τι θέλουμε να αφαιρέσουμε εμείς και πρέπει μετά να δούμε τι θα απομείνει αφού βγάλουμε αυτό και εκείνο. Και αυτή είναι πραγματικά η ισορροπημένη πρόταση που χρειαζόμαστε για τη σύγχρονη αγορά τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε να διατηρήσουμε και την διεθνή ανταγωνιστικότητά μας. Uh, full quality of um, Συμμερίζομαι τις ανησυχίες όλων για την ε, υψηλή ποιότητα ε, και το, τωρινό πακέτο τηλεπικοινωνιών η σχετική οδηγία τώρα υλοποιείται στα κράτη-μέλη, τώρα εφαρμόζεται ή πολύ πρόσφατα εφαρμόστηκε. Δεν έχουμε λοιπόν feedback, δεν έχουμε στοιχεία. Ε, τούτου λεχθέτως ε, ας περάσουμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Εγώ καλωσορίζω τα μέτρα που είναι φιλικά προς τον καταναλωτή και προς τον ανταγωνισμό, αλλά θα πρέπει να δούμε τι αξία μπορούμε να προσθέσουμε και εμείς, τι μπορούμε να συνεισφέρουμε. Νομίζω ότι πρέπει να περιοριστούμε ε, το να δώσουμε την γνώμη μας, την άποψή μας, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι Λαμβάνεται υπόψη η γνώμη μας. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για το φάσμα, για τον συντονισμό, για τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του ραδιοφάσματος, το άρθρο 23 για το δωρεάν και ανοιχτό διαδίκτυο, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας των δεδομένων, για τα εχέγγυα, για την ποιότητα των δεδομένων. Ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδίου κειμένου της ε, Κομισιόν είναι η ουδετερότητα του δικτύου. Αλλά η έννοια αυτή ε, δεν έχει κάποιο νομικό ορισμό. Ε, επίσης, τι σημαίνει η διαχείριση της ε, διακίνησης των στοιχείων. Και τι σημαίνει η πρόσβαση στις ε, ε, υπηρεσίες και στις εφαρμογές μέσω διαδικτύου. Για τη διαχείριση του φάσματος. Νομίζω πολύ σημαντική είναι η πληστηριασμή ραδιοσυχνοτήτων. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν ε, έντονα σε αυτό. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, δύσκολο θέμα συζήτησης με το Συμβούλιο, το οποίο θέλει να κρατήσει τον έλεγχο στον τομέα, νομίζω ότι καλό είναι να υπάρξει καλύτερος, καλύτερος συντονισμός και ανταλλαγή κοινών εμπειριών για τους πληστηριασμούς του φάσματος. Η Κομισιόν ήδη έχει επεκτείνει τις αρμοδιότητες συντονισμού του φάσματος Ίσως οι αρμοδιότητες αυτές δεν είναι αρκετά εκτεταμένες ή αρκετά αποτελεσματικές. Ίσως να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική χρήση των αρμοδιοτήτων που ήδη διαθέτουμε πριν τις επεκτείνουμε. Εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για την χρήση αυτών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα και ελπίζω να σημειωθεί πρόοδο στο σημαντικό αυτό θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Doris. Και ευχαριστώ την Πέτρα για αυτή την παρουσίαση που μας έκανε και θα ξεκινήσω με αυτό που το στο τέλος, ότι ε, δεν είναι πολύ καλή η σύνταξη αυτού του κειμένου και το καλύτερο συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε είναι να αποσύρει την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά αυτό μπορεί να μην συμβεί αλλά θα ήταν καλό αν μπορούσαν να το κάνουν ναι, κάτι τέτοιο. Θέλουμε να έχουμε ανοιχτά δίκτυα, να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση στις πληροφορίες και πρέπει και η Ήτρε να είναι ξεκάθαρη προς αυτό. Πρέπει να ε, το υποστηρίξουμε αυτό, για ε, ε, να είναι δημόσιο αγαθό οι συχνότητες φάσματος και να δούμε και ποιος, ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος στην πολιτισμική ζωή πρέπει και αυτό να φανεί και αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι αρκετά σαφές στο έγγραφο της Επιτροπής. Και το ίδιο ισχύει και για τις βέλτιστες προσπάθειες, την αρχή των, της βέλτιστης προσπάθειας. Και επίσης για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες πρέπει να διαχωρίσουμε το πρωτόκολλο του διαδικτύου και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε διάφορα παραδείγματα για αυτές τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αυτό το είπε και η Σαμπίνα. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτές δεν είναι ειδικέ υπηρεσίες. Ε, συνήθως ε, είναι διαθέσιμες και μέσω του κανονικού διαδικτύου. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε αυτό τον όρο. Η κυρία Μίχελς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα και σας ευχαριστώ για την ισορροπία με την οποία παρουσιάσατε αυτή την έκθεση, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπατε και με τις τροπολογίες και γι' αυτό δεν χρειάζεται να υποβάλουμε άλλε τροπολογίε. Από την πλευρά τη δική μα Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να καλύψουμε και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό, δηλαδή την πολυμορφία των δικτύων και ότι οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες. Ε, σε όλους και αυτό μας φαίνει σε έναν κοινό στόχο. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε εμείς ως Επιτροπή. Και αυτό μας επαναφέρει και στις συζητήσεις που είχαμε σήμερα το πρωί, όταν είδαμε την ε, πράσινη βίβλο. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου σωστός τρόπος αυτός για να προχωρήσουμε αυτό που μας λέει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε εμείς να υπερασπιστούμε τον ανοιχτό χαρακτήρα και όχι να το αμφισβατήσουμε αυτό. Μιλάνε για ευρυζωνικότητα και την ίδια στιγμή έρχονται και προτείνουν κάτι τέτοιο όπως αυτός ο κανονισμός. Δεν μπορούμε να, να συμφωνήσουμε με μια τέτοια κατεύθυνση γιατί αυτό δεν βασίζεται ουσιαστικά στην πραγματική δημοκρατία. το λογικό θα ήταν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει αυτό, αυτή τη νομική πρόταση. Και δεν ξέρω τι θα πούνε και οι άλλες επιτροπές, αλλά ίσως μετά μπορούμε να στείλουμε ξανά ε, τις προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τις πούμε ότι αυτό δεν είναι πραγματική ουσιαστική δημοκρατία. αυτό είναι σίγουρα ένα ε, ε, παράδειγμα κακής ε, επίδοσης από την πλευρά των θεσμών. Ε, επαναλαμβάνω λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, συμμερίζομαι τις απόψεις σας. Η κυρία Σακ, ευχαριστώ. Ήδη αρκετά υπόθηκαν για αυτή την πρόταση για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Πρέπει να δούμε και ποια είναι η φιλοδοξία πίσω από αυτή την πρόταση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν ε, να σταματήσει αυτό το υπερβολικό κόστος ε, περιεγωγής που και έχουμε και τις ευρωεκλογέ μπροστά μας και πρέπει να εστιάσουμε στο πεδίο εφαρμογή που έχει η δική μας Επιτροπή και νομίζω ότι πρέπει να ε, επικεντρωθούμε στο δημόσιο συμφέρον που έχει αυτό. Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με την πρόσβαση στην ενημέρωση και αυτά είναι ε, παιδί, ε, με το οποίο ασχολείται η Επιτροπή μας. Σε πολλά σημεία η πρόταση δεν είναι σαφής και πολλές φορές το Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ της ουδετερότητας ε, και της πολυμορφίας και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να βασιστούμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιστροπής υπάρχουν ε, προτάσεις ε, που λένε ότι ε, αναφέρονται στην διαδικτυακή ουδετερότητα, αλλά ουσιαστικά δεν είναι διαδικτυακή ουδετερότητα ή τουλάχιστον εμείς δεν το καταλαβαίνουμε έτσι. Για το ανοιχτό διαδίκτυο πρέπει να επιτρέπουμε να υπάρχει χώρος για τις επιχειρήσεις να έχουν και να μην επιτρέπουμε να υποβαθμιστεί η καινοτομία από τις ε, επιχειρήσεις ε, startup, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και τους ε, καταναλωτές. Και μετά πρόσβαση στον πολιτισμό, πρόσβαση στη γνώση και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε στους μεγάλους παίκτες της αγοράς, πρέπει να είναι ένα δημόσιο αγαθό, μια δημόσια αξία. Συμφωνώ λοιπόν και με ε, αυτό που είπε η κυρία Πάκο, ότι πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες. και να είναι σταφείς οι ορισμοί όσον αφορά και την ποιότητα των υπηρεσιών και για το φάσμα τώρα η ομάδα μας είναι υπέρ της εναρμόνισης για τους στόχους της ε, ενιαίας αγοράς, να χρησιμοποιήσουμε ε, αγορά ε, γιατί το διαδίκτυο θα είναι σημαντικό και για την, για την τηλεόραση. Πρέπει να δούμε πώς έχει πραγματικότητα τώρα και να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι, οι προτάσεις για το φάσμα και για την ουδετερότητα και να είναι χρήσιμες και για το μέλλον να δούμε ποιος είναι ο ρόλος μας ως νομοθέτες, όχι να ε, ε, ρυθμίσουμε υπερβολικά, αλλά να προστατεύσουμε κάποιες αρχές και να προστατεύσουμε τις αρχές της, του ανταγωνισμού, της πρόσβασης στον πολιτισμό και στην γνώση, ε, την καινοτομία. Και αυτά είναι τα στοιχεία που ήθελα να αναφέρω εγώ για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας στραφούμε στην Κομισιόν να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Um, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Την άκουσα με άκρα προσοχή. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Νομίζω έγινε μια αναφορά στο σχεδόν πλαίσιο την επιλογή, μάλλον την εφαρμογή του και γιατί αφού είναι λυπής ακόμη έρχεται με νέες προτάσεις η Κομισιόν. Καταρχάς, αληθεύει ότι το ισχύον πλαίσιο άρχισε να εφαρμόζεται από το 2011 και καθυστέρησε σε πολλές περιπτώσεις ε, η μεταφορά του στο εθνικό δίκαιο. Και υπάρχουν μελέτες για το πώς εφαρμόζεται, τι ε, ποσοστά εφαρμογής ε, και μεταφοράς έχουμε και θα σας πω ε, καταρχάς ότι αυτά τα ενδικά μέσα, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τι μέσα δηλαδή χρησιμοποιούν όταν ρυθμίζουν τα σχετικά. Μελέτη αντικτύπου. Ασκήθηκε κριτική. Αν δείτε πολύ προσεκτικά το παράδειγμα 1 2, θα δείτε ότι δίνει ξεκάθαρα παραδείγματα ρυθμιστικών αποφάσεων από τις ρυθμιστικές αρχές και το ισχύον πλαίσιο Ουσιαστικά μιλάμε για μεγάλη ποικιλία, αν θέλετε, στην εφαρμογή των ρυθμίσεων. Σίγουρα δεν είναι επαρκές στο πλαίσιο, χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό σίγουρα και για την Επιτροπή σας είναι το ανοιχτό δίκτυο και η ιδιαιτερότητα του δίκτυου. Γιατί τώρα να προβούμε σε ρύθμιση. Και γιατί θεωρούμε ότι έχουμε σαφή παραδείγματα και στην προκειμένη περίπτωση που δείχνουν ότι υπήρξε αποκλίνου, υπήρξαν αποκλίνουσες προσεγγίσεις από τα κράτη-μέλη. Σε δύο κράτη-μέλη υπάρχει νομοθεσία περιουδετερότητας. Σε κάποια άλλα λίγα κράτη-μέλη, η αρχή δραστηριοποιήθηκε και στον έλεγχο και στην έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών. Αλλά υπάρχουν κράτη-μέλη αρκετά όπου ο αριθμιστικός φορέας δεν έλαβε κανένα μέτρο σε ό,τι αφορά την ουδετερότητα του δικτύου. Βέβαια, αν δει κανείς ε, τις έρευνες ε, της Μπέρεκ για την κίνηση ε, στο διαδίκτυο λίγο χρόνια πριν, το 12 δόθηκαν στη δημοσιοτήτα τα πορίσματα, έδειξαν ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και οι δημόσιες διαβουλεύσεις, δύο τον αριθμό, για την δικτυακή ουδετερότητα έδειξαν ότι υπάρχουν προβλήματα. Άρα νομίζουμε ότι μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε για το ότι χρειάζεται ε, να υπάρξει αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε τον έλθω στην ουσία. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε εύκολα να συμφωνήσουμε μαζί σας Ω προ τι αρχέ που ακούστηκαν και σε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή ανάγκη εξασφάλιση ενό ανοιχτού διαδικτύου. Οι καταναλωτέ, οι τελικοί χρήστε θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πληροφορίε και στο περιεχόμενο και σε εφαρμογές, ένα ανοιχτό διαδίκτυο από τη μία και από την άλλη πλευρά οι πάροχοι περιεχομένου και εφαρμογών να έχουν τη δυνατότητα να έχουν χώρο για καινοτόμες νέες υπηρεσίες. Και αυτός ακριβώς είναι και ο δικό μας στόχος με την πρόταση που υποβάλλουμε. Έπειτα, υπάρχει το ζήτημα των εξειδικευμένων υπηρεσιών. Συνόγω από τη συζήτηση ότι επί της ουσίας δεν διαφωνείτε. Νομίζω ότι είναι ευρέως ε, αποδεκτό ότι και τώρα, αλλά δηλαδή, ιδίως στο μέλλον, θα πρέπει να μπορούμε να εγγυηθούμε μια δεδομένη ποιότητα για τις υπηρεσίες που παρέχουμε, για νέες εφαρμογές, ιατρικές υπηρεσίες, παρακολούθηση ιατρικών υπηρεσιών ήταν ένα παράδειγμα. αλλά και στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη της καινοτομίας. Τώρα μπορούν να συμβιώσουν αυτά τα δύο. Αυτός είναι ο στόχος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σοβαρά αντιμετωπίζει το θέμα. Γι' αυτό και έχουμε εισαγάγει ασφαλιστικέ δικλείδε στην πρότασή μα, τουλάχιστον κατά την άποψή μα. Αυτέ θα εγγυώνται το άνοιγμα του διαδικτύου. Υπάρχουν απαιτήσει για τους παρόχους ε, του πρωτοκόλλου του διαδικτύου ISPs, όταν παρέχουν μια εξειδικευμένη υπηρεσία, η ποιότητα της ε, υπηρεσίας προς το διαδίκτυο να μην ε, αποδυναμώνεται να μην υποβάθμιζετε ώστε να τίθεται σε κίνδυνο ευέλιστη προσπάθεια. Κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε, θα πρέπει να έχουμε εχέγγυα για τους τελικούς χρήστες όταν να σε επαφή με τους ε, παρόχους των διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε να ξέρουν ακριβώς ε, σε τι υπηρεσίες ε, συγκατατίθενται. θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες για την ταχύτητα και αν δεν ε, εφαρμόζονται οι όροι των συμβάσεων, θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε λοιπόν πάλι ασφαλιστικέ δικλείδε που εγγυώνται το ανοιχτό χαρακτήρα του διαδικτύου. Έπειτα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πώ θα πρέπει να οριστεί, να εντοπιστεί, βέλτιστη προσπάθεια, ποια είναι η τεχνολογία που μπορεί να παρέχεται από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ή αν θα πρέπει να ορίσουμε τις τεχνολογίες ή τις τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πάροχοι των διαδικτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση της κίνησης στο διαδίκτυο. Η Κομισιόν θεωρεί ότι εάν θέλουμε να έχουμε έναν κανονισμό που θα μπορεί να ισχύει και στο μέλλον, δεν θα πρέπει να είμαστε... Δεν θα πρέπει να φέρουμε τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, γιατί θα μπορεί μετά να εφαρμοστεί ο κανονισμός άπαξ και εγκριθεί, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Ίσως να σταματήσω εδώ για την ε, ουδετερότητα και μετά να μιλήσω για το φάσμα. Λίγα λόγια μόνο. Στηρίζουμε και εμεί την ανάγκη να υπάρχει μια συντονισμένη προσέγγιση για το φάσμα και για την ζωνικότητα και για το πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Είναι σημαντικό το φάσμα και η στόχη της δημόσιας πολιτικής για τις γενικές υπηρεσίες, προώθηση πολυγλωσσίας, πολιτισμικής ποικιλομορφής κτλ νομίζω ότι δεν θίγονται αυτοί οι στόχοι με τον προτινόμενο κανονισμό. Και κάποια άλλα σημεία. Η πρόταση δεν προκαταλαμβάνει πολιτικές αποφάσεις για την εναρμόνιση του φάσματος για την ασύρμετευρυζωνικότητα. Οι διατάξεις που έχουμε στον προτινόμενο κανονισμό εφαρμόζονται μόνον αφού υπάρξει η εναρμόνιση του φάσματος για την ασύρματη ευρυζωνικότητα. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Μόνο το ενεργοσμένο φάσμα για ευρυζωνικότητα αποτελεί το της πρότασης, άρα το φάσμα για τους ραδιοτηλεπτικούς φορείς δεν περιλαμβάνεται. Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Αυτά θα καθοριστούν και οι προθεσμίες μόνο μετά την αρμόνιση του φάσματος για την ασύρματη ευρυζωνικότητα. Uh, Υπήρξε και ένα ερώτημα για τον ισχύοντα συντονιστικό μηχανισμό. Αφού δεν... Γιατί χρειαζόμαστε κάτι νέο, κάτι πιο ισχυρό. Οι διαδικασίες απόδοσης φάσματος δεν αποτελούν αντικείμενο ουσιαστικά καθόλου ε, συντονισμού μέσα στο ισχυρό πλαίσιο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι με αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. ή αν θέλετε περιττέρω εναρμόνιση, περαιτέρω συντονισμό. Και σταματώ με αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η εξυπνάδα μου διατηρείται αμύωτη αλλά πραγματικά δεν μπορώ να δω... Δεν βλέπω να έχουν δοθεί απαντήσεις στις ερωτήσεις που έγιναν. Ας είμαστε ανοιχτοί. Ε, έχουμε πολλά που έχουν συμβεί στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Ε, δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας για το τι έχει συμβεί στις τηλεπικοινωνίες, γιατί αν δεν κάνουμε εμείς κάτι, θα αναλάβουν άλλοι. Δεν νομίζω ότι η πολιτική ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για κάτι άλλο. Ε, δεδομένης της κατάστασης των πραγμάτων, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο χρησιμοποιείται τα 800 αυτά δίκτυα πριν ολοκληρωθεί ε, αυτή η άσκηση ελέγχου που, κάνουν, που κάνουμε. Ε, πρέπει μέχρι ε, το 2015 να δούμε πώς έχει η κατάσταση και αν είναι 800 ή 700. Και πολύ φοβάμαι ότι η Επιτροπή δεν κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πολλές φορές σταματήσει στα 700 τα τελευταία χρόνια. Ξέρω ότι ε, ε, Ξέρω, για παράδειγμα, στην εκλογική μου περιφέρεια, τα θέατρα, για παράδειγμα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ε, αμοιβέ και στις χρεώσεις δεν ξέρω αν ένα ταμείο για τις τηλεπικοινωνίες ε, θα ήταν ε, η σωστή λύση. Τώρα μας λένε ότι τα κράτη πρέπει να το αναλάβουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το αναλάβει το κράτος. Ε, και να πρέπει το θέατρό μου να αλλάξει γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση της ε, Κομισιόν και το καλύτερο θα ήταν από την πλευρά σας να αποσύρετε αυτή την πρόταση. Γι' αυτό και συμφωνώ με αυτά που είπαν ε, οι συνάδελφοι. Ε, υπάρχουν και άλλες επιτροπές που δεν συμφωνούν με την πρότασή σας και δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό να γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Πέτρα, θέλεις και εσύ να ανταποκριθείς σε αυτά που είπε η Κομισιόν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπες, Ντόρις. Συμφωνώ πλήρως. Εν τέλει, δεν μας δόθηκαν απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάναμε. Δεν λάβαμε απαντήσεις. Μοιάζει να υπάρχει ένα μόνιμο παραπέτασμα καπνού ε, ενδιαφέρον έχει ότι όταν κάνουμε λόγο για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εκείνοι μας λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει το ψηφιακό έλλειμμα, ότι δεν τους ενδιαφέρει η χρήση αυτού του εύρους ζώνης, γιατί καλά τα πάμε όπως είμαστε τώρα και όλη η συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό των κρατών μελών για τη χρήση των συχνοτήτων Πρέπει να δούμε τι λύσεις δίνουν τα κράτη-μέλη πρώτα απ' όλα και να δούμε εάν θα αποφασίσουν, ε, πώς θα αποφασίσουν να μοιράσουν την πίτα στο μέλλον. Ε, ε, μεταξύ ραδιοτηλεπτικών σταθμών, παραγωγών πολιτισμικού περιεχομένου. υπάρχουν διάφορα λόμπι που κάνουν τη δουλειά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει εμείς να ορίσουμε πράγματα που άλλοι είναι πιο αρμόδιοι να ορίσουν. Τώρα για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η Μαρίκα επίσης ε, εξέφρασε τα ίδια επιχειρήματα. Αν ε, είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι το κείμενο της Κομισιόν δεν μας λέει τι είναι εξειδικευμένες υπηρεσίες. Και αν ρωτήσεις τον κόσμο, ε, ακούς IPTV και απορώ πως αυτό συνδέεται με τις εξειδικευμένες ε, ε, υπηρεσίες. Και απ' την άλλη υπάρχει το e-hills, δεν ξέρω και αυτό τι σχέση έχει με τις... Α, η, με συγχωρείτε, η ηλεκτρονική υγεία, το e-health. Ακούμε και αυτό να ορίζεται ως περιεχόμενο των ε, εξειδικευμένων υπηρεσιών. Was ansonsten Anwendungsbereiche angeht, habe ich bisher keine... Άλλες χρήσεις υπάρχουν. Δεν έχω λάβει απαντήσεις. Αν δει κανείς τον εξειδικευμένο τύπο, την εξειδικευμένη λογοτεχνία, τις λεγόμενες managed services, τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες ή τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εναλλάξ. Στην πραγματικότητα είναι υποσυστήματα του διαδικτύου που μπορούν να συμπεριληφθούν σε πακέτα. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να πούμε πως υπάρχουν πακέτα που θα υποκαταστήσουν το ελεύθερο και ανοιχτό διαδίκτυο. Εμείς δεν, θέλουμε αυτό να κάνουν, ε, ε, δεν θέλουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες να κάνουν αυτό και ούτε χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ε, αν μπορεί κάποιος να το πει με μεγαλύτερη σαφήνεια από μένα, παρακαλώ πέστε το. Έχουμε αυτόν τον ορισμό των εξειδικευμένων υπηρεσιών τον οποίο τον άλλαξαν κιόλα και λένε πως είναι ε, υπηρεσίες ηλεκτρονικές σε κλειστό κύκλωμα ε, ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο του διαδικτύου. Δεν είναι υποσύστημα λοιπόν του διαδικτύου και δεν αντικαθιστούν κομμάτια του δικτύου, ούτε χρησιμοποιούνται προς αντικατάσταση τμήματων του διαδικτύου. Αυτός είναι ο μόνος ορισμός που είδα για, τον, ε, την οριοθέτηση του τι είναι αυτές οι εξειδικευμένες υπηρεσίες. Ε, θέλ, χρειαζόμαστε έναν ορισμό. Ε, αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερόμενων. Για παράδειγμα, το κύκλωμα της ηλεκτρονικής υγείας, το e-health, η δικτύωση των νοσοκομείων, τα επιχειρηματικά μοντέλα, B2B, αυτά δεν πρέπει να τα βλέπουμε ως ξεχωριστά δίκτυα σε σχέση με το κλασικό διαδίκτυο. Κανείς δεν μου έχει εξηγήσει σωστά τι είναι αυτές οι εξειδικευμένες υπηρεσίες. Εγώ προσπάθησα να τις ορίσω η ίδια. Πράγμα ε, πάντως δεν είναι το σύνηθες ίντερνετ. Εάν κάποιος γνωρίζει καλύτερα από μένα, παρακαλώ να το πει για την ουδετερότητα. Πάντοτε τη ζητούσαμε, ε, η κυρία Κρούς ε, ε, ήταν παρούσα κατά την πρώτη ακρόαση και κατά την πρώτη ανάγνωση. Η κυρία Κρούς τόνισε τη σημασία της δικτυακής ουδετερότητας Όταν πρώτο, είπαμε ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η ουδετερότητα όποια άποψη και αν υιοθετήσουμε για την, το περιεχόμενο αυτής της ουδετερότητας. Πολλές φορές ρωτήσαμε την Επιτροπή και πάντοτε μας απαντούσε δεν είμαστε ακόμα σίγουροι υπάρχει αυτό το φράγμα, αυτό το εμπόδιο μεταξύ μας και ξαφνικά έξι μήνες πριν από τις ευρωεκλογές βγαίνει αυτή η έκθεση, αυτό το σχέδιο κανονισμού και ξαφνικά πρέπει να επιταχύνουμε ε, το, το, το Κοινοβούλιο έχει προσπαθήσει να το περάσει αυτό τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Προσπαθήσαμε να υπάρξει μια σωστή και λογική έκθεση, ένα καλό πακέτο για την ουδετερότητα και τώρα τι γίνεται, ε, έρχεται το, το, το Σεπτέμβριο και πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε να κάνουμε κάτι. Πολύ φοβάμαι ότι έχουν ε, από πίσω υποκρύπτονται κάποιες ε, ανίερες συμφωνίες, τις οποίες δεν είμαι καθόλου διατεθειμένη να στηρίξω και να προάγω. Και δεν πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε αυτό. Όσο αφορά τις ε, προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις και τις αγροτικές περιοχές ε, και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες έχουν θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ε, σε επικαιροποιημένο, ενημερωμένο δίκτυο. Αν δείτε τις αγροτικές περιοχές, Αν δείτε το χρόνο, την, την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων σε αγροτικές περιοχές, ε, είναι το ένα δέκατο, το 1, το εικοστό, το ένα χιλιοστό της ταχύτητας των πόλεων. Οπότε λέμε ναι, υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε αγροτικές περιοχές, αλλά είναι τόσο αργή αυτή η πρόσβαση που τελικά κανείς δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και το είπα και πολύ ξεκάθαρα και αυτό ότι η σύνθεση με το διαδίκτυο πρέπει να πληρεί κάποια, κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ε, και πρέπει τεχνικά να είναι επικαιροποιημένο το σύστημα, να είναι σύγχρονο και πρέπει αυτό να ενταχθεί στις ε, αντίστοιχες συμβάσεις. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ο Μάλκον Χάρβερ όταν μιλούσε για τις απαιτήσει διαφάνειας σε πολλές παραγράφους ε, καλά όλα αυτά, αλλά δεν είναι νομοθετημένο αυτό, οι απαιτήσει διαφάνειας. Βασικά το λογικό είναι να κατανοεί κανείς τι είναι γραμμένο στη σύμβαση, ποιοι είναι οι συμβατικοί όροι. Υπάρχει αυτή η προϋπόθεση και η απέτηση εξασφάλισης ενός κατώταρου, κατώτε του ορίου. Αλλά πολύ συχνά, όπως ανέφερα, στις αγροτικές περιοχές δεν πληρούνται αυτές οι προδιαγραφές. Σκέφτηκα ε, να προτείνω στην Επιτροπή μας απλά να απορρίψουμε αυτήν την έκθεση. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει πλειοψηφία στην, στους κόλπους της Επιτροπής για κάτι τέτοιο. Αλλά δυστυχώς οι άλλες δύο Επιτροπές ε, αμέριμνα συνέχισαν να ασχολούνται με το θέμα. Και δεν μπορέσαμε να έχουμε έτσι μια, ένα κοινό μέτωπο. Ε, αν πάλι εμείς το απορρίπταμε, δεν θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε στο παιχνίδι θα αποκλειόμασταν τελείως από κάθε συζήτηση. Πάντως, εάν το απο... τεχνικά θα ήταν πιο ορθό να πούμε, ας προσπαθούμε να το βελτιώσουμε το κείμενο αυτό, αντί να το απορρίψουμε. Δεν πρέπει πάντως να το μετακυλήσουμε την ευθύνη στο επόμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνω τη συζήτηση για αυτό το θέμα. 5 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η πρόσθεση μία για τις τροπολογίες, όχι αυτό που έχετε στα εγγραφά σας, 5 Δεκεμβρίου, γιατί χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο. 5 Δεκεμβρίου λοιπόν. Υπάρχουν αντιρρήσεις? αν όχι λοιπόν κρατάμε το 5 Δεκεμβρίου για την προθεσμία Πέτρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, ευχαριστώ και την Κομισιόν. Και τώρα περνάμε στο σημείο 9 της σημερινής διάταξης. Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν κόσμο με πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές. Ο κύριος Παπανικολάου είναι εδώ έχει καταρτήσει ένα σχέδιο γνωμοδότησης για αυτή την έκθεση για την εξωτερική πολιτική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν κόσμο στον οποίο επικρατούν πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές. Yeah. Thank Ελπίζω ότι αυτό το θέμα δεν θα είναι τόσο δύσκολο όσο το προηγούμενο. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο γνωμοδότησης που με χαρά σας παρουσιάζω εδώ σήμερα ε, αναφέρεται και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και είναι σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν κόσμο με πολιτισμική και θρησκευτικές διαφορές. Είναι μια γνωμοδότηση ιδίου πρωτοβουλίας, αλλά είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολιτισμική και σέφεται τις ε, ε, παραδόσεις και αυτό φέρνει την προστιθεμένη αξία στις πολιτικές μας. Χρειαζόμαστε αηφόρο ανάπτυξη η ειρήνη και διάλογο μεταξύ των ε, πολιτισμικών. Αυτές οι αρχές αποτελούν μέρος της ε, Σύμβασης UNESCO 2020 για την προστασία των πολιτισμών και σε αυτό αναφερόμαστε επίσης στο σχέδιο ε, γνωμοδοτησής μας. Η μορφία συμπεριλαμβάνεται και στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία είχαμε υιοθετήσει στην τελευταία Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Πρέπει να προωθήσουμε την πολυμορφία και τον θρησκευτικό διάλογο, να είμαστε κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, κατά του φανταμετρισμού, να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, να είμαστε κατά της ε, ε, βίας με την εμπλοκή όλων των φορέων και άλλων χωρών, τρίτων χωρών, μπορούμε να έχουμε καλύτερες πρωτοβουλίες στην κατάρτιση των νέων, στην ε, πολυγλωσία, στα αθλήματα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εξωτερικές σχέσεις. Μπορούμε να επενδύσουμε στις γνώσεις, στο να γνωρίσει κανείς καλύτερα τους άλλους πολιτισμούς Πρέπει να υπογραμμίσουμε επίση ε, και τα ξένα μέσα μαζική ενημέρωση. Κάθε φορά που έχω την ευκαιρία το κάνω αυτό. Μιλάω για τα ξένα μαζική ενημέρωση ε, γιατί ε, μα δίνει μια πρόσβαση σε άλλα πολιτισμικά αγαθά. Και επίση είναι σημαντικά δίκτυα όπω το Ευρωπαϊκό. Η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιεί την πολιτισμική διπλωματία και αυτό είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο που έχουμε για την εξωτερική πολιτική και θα βελτιώσει τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι πριν από κάποιες δεκαετίες ο Μονέ, ο Ζαμονέ, είχε πει ότι αν έπρεπε να ξαναξεκινήσει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα την ξεκινούσε με τον πολιτισμό η αρμοδιότητα της Επιτροπής μας σε αυτό το θέμα είναι περιορισμένη. Προσπαθήσαμε λοιπόν να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο κείμενο που να ε, ορίζει αυτά που θέλουμε, τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε και τώρα ανυπομονώ να ακούσω τις ε, απόψεις σας και με χαρά να δουλέψω πάνω στις ε, τροπολογίες σας και περιμένουμε όλες τις προτάσεις σας και τις ιδέες σας ε, ό,τι ιδέες έχετε για τροπολογίες, συνεισφορές γενικότερα. Ευχαριστώ τη γραμματεία, την κυρία Έριξον. Ευχαριστώ επίσης ε, τον Σάντος και τον σύμβουλο ε, Ρομπέρτο Γιανέλα. Και σας ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων για τα σχόλιά σας και τις συνεισφορές σας και ελπίζω ότι δεν μακρηγόρησα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Ευχαριστώ. Τώρα δυστυχώς θα ε, εκπροσωπήσω ότι είναι μία, είναι δύσκολη δουλειά αυτή, είναι σκιώδης η συγγήτρια. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για, αυτή, για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Πρώτα απ' όλα, για τις σχέσεις ε, με τις ε, τρίτες χώρες. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο πολιτισμός είναι όντως ένα εργαλείο για την, για την εξωτερική πολιτική και πρέπει να το χρησιμοποιούμε περισσότερο αυτό το εργαλείο, περισσότερο από ό,τι το έχουμε χρησιμοποιήσει έως τώρα. Και νομίζω ότι είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι παραπάνω από μια οικονομική ζώνη, από μια οικονομική δύναμη. Είναι ένα πολιτισμικό και πολιτικό σχέδιο. Και αυτό πρέπει, αυτή πρέπει να είναι η εικόνα που θα δίνουμε στον κόσμο. Πρέπει να έχουμε τέτοιες ε, εταιρικές σχέσεις πολιτισμικές και πολιτικές με τις άλλες χώρες. Ε, το πολιτισμικό συστατικό στοιχείο, η, η, η Εμίλια θέλει να είναι ακόμα πιο ορατό. να, να πούμε ότι στηρίζουμε την ε, ποικιλία των ε, πολιτισμών και νομίζουμε ότι έτσι θα ήταν σαφέστερο το μήνυμα για τις τρίτες ε, χώρες. Να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο για τον πολιτισμό και να συμπεριληφθεί στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως κάποιες θεμελιώδεις αρχές για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες να συμπληρώνουμε έτσι δηλαδή τις δράσεις που λαμβάνουν, αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Να, να υπάρχει σαφής εντολή για να παρουσιάζεται κάθε φορά η πολιτιστική κληρονομιά και να γίνεται ορατή σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενισχύσουμε μόνο τους οικονομικούς δεσμούς που έχουμε με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και τους πολιτισμικούς δεσμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την πολιτισμική συνεργασία με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ενισχύσει την εικόνα της και της Ένωσης και των ε, μελών της και να βελτιώσει την ε, πρόσβαση ε, στις αγορές πολιτισμικών αγαθών. Έτσι θα αυξηθεί και η προσωπική επαφή, η προσωπική επαφή μεταξύ των ανθρώπων και Φυσικά αυτά είναι στοιχεία τα οποία ε, ε, στηρίζουμε απόλυτα. Χαιρετίζουμε λοιπόν ε, και τις προσπάθειες που έχουν γίνει ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Να πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τον κόσμο, αλλά να πούμε και ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές αξίες και όχι απλά να αποδοκιμάζουμε, αλλά να κάνουμε προσπάθειες για να συνδεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ. Κοριάν, πρώτα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλά κάναμε ε, και εκδώσαμε μια γνωμοδότηση για αυτήν την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων γιατί, εντάξει βέβαια πολλά υπολείπονται σχετικά με την εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική. Σίγουρα είχαμε περισσότερες προσδοκίες ε, από αυτόν τον τομέα, από αυτή την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πολύ φοβάμαι ότι στήσαμε ένα μεγάλο οικοδόμημα κενό νοήματος στο εσωτερικό του. Εν περιπτώσει. Σε σχέση με αυτά που παρουσίασε ο συνάδελφος ε, Παπα-Νικολάου ε, και το soft power, όπως είπε η κυρία Κάμεμπερτ, ε, προσπαθούν να δώσουν λίγο περισσότερη ουσία στις εξωτερικές σχέσεις στον τομέα του πολιτισμού. Ε, πρέπει να έχουμε εργαλεία και μέσα στη διάθεσή μας, αν θέλουμε να δώσουμε αυτή τη διάσταση στην εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική. Μια ενότητα, ένα κοινό πλαίσιο πάνω απ' όλα, ε, που να σέβεται τις ε, τοπικές ιδιαιτερότητες και διαφορές και να αγκαλιάζει τους πολίτες, τη δημιουργικότητα, ε, στις εξωτερικές σχέσεις. Νομίζω ότι πρέπει το βάρος, ε, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στον πολιτισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Σκάκη, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βλέπω την γνωμοδότηση αυτή γιατί πραγματικά έχει να κάνει και με δουλειά που έκανα εγώ προηγουμένως στην Επιτροπή μας, σε συνεργασία με όλου εσά, όταν εξετάζαμε την πολιτισμική συνιστόσα τη ε, εξωτερική πολιτικής τη Ένωση και πολλά από αυτά που αναφέρατε είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ θετικές ε, υποδείξεις. Η αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να παίξουν νέε τεχνολογίες, ε, διασύνδεση ανθρώπων στο περιεχόμενο από όλο τον κόσμο, φυσικά δεν θα σα εκπλήξω ότι είμαι υπέρ Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο των νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση του διαπολιτισμικού ή διαθρησκευτικού διαλόγου, να μην τον περιορίσουμε μόνο εκεί, γιατί πολλά άλλα μπορούν να κάνουν οι νέε τεχνολογίε. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την ελευθερία στην Ευρώπη, ώστε μπορούμε όλοι μα να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό. Θα πρότεινα λοιπόν να μην τους πούμε ε, τι να κάνουν, αλλά να τους εκφράσουμε τις αξίες που εκπροσωπούνται και μέσω της πολιτισμικής αυτής ποικιλομορφία, ε, που δείχνουν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει περιορισμός και γι' αυτό η Ευρώπη είναι μοναδική. Δηλαδή να μην είμαστε, ε, να μην προβαίνουμε σε υπαγορεύσεις πιο πολύ αν θέλετε, να είμαστε πιο ανοιχτοί. Γιατί μπορούμε έτσι να δώσουμε ένα πολύ πιο ηχηρό μήνυμα και να παρουσιάσουμε ε, τι πιστεύουμε ότι είναι αυτό που μας κάνει περήφανος για την Ευρώπη και την πολιτισμική της ποικιλομορφία. Φύσα, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο Λαου για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν. Τόσες, ε, σε τόσες χώρες εκπροσωπούνται, σε τόσες χώρες έχουμε πρέσβεις που θα έπρεπε να προωθούν την ε, ευρωπαϊκή πολιτισμική και πολιτιστική ποικιλομορφία. Εάν, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, έχουμε κάτι για το οποίο μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι στην Ευρώπη, είναι ο πολιτισμός μας, η πολιτισμική πολυμορφία, η πολυγλωσία, ο πλούτος ε, των γλωσσών των ευρωπαϊκών και πρέπει να τα προβάλλουμε αυτά που αποτελούν ε, πλέον εκτήματα δικά μας που δεν τα έχουν άλλες ε, ήπειροι, άλλες χώρες και αυτό είναι και καθήκον των πρεσβευτών θα πρέπει επίσης ε, να μιλήσουμε και για τον τουρισμό και για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την προώθηση ε, των διαφόρων πολιτιστικών φεστιβάλ, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ε, οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύσεις κτλ. Όλα αυτά θα βοηθήσουν και τον τουρισμό και την οικονομία. Και παραλαμβάνω ότι πρέπει να επιφορτιστούμε το καθήκον αυτό και οι ξένοι οι πρεσβευτές μας στις ξένες χώρες. Θα ήθελα να σας πω ότι ακριβώς τώρα έχουμε και τη... το βραβείο Λουξ. Θα ξεκινήσει η τελετή. περσινή νικήτρα, When She Άννα Κέλλερ, θα τη θυμάστε, ένα τέτοιο παράδειγμα θα ήταν καλό. Μέχρι και στο Πακιστάν προβλήθηκε αυτή η ταινία. Γιατί και το θέμα και εκεί είναι κάτι που ενδιαφέρει. Πρέπει λοιπόν πράγματι να αξιοποιήσουν οι αντιπροσωπείες μας οι εκπρόσωποι, οι ακόλουθοι των εξωτερικών υποθέσεων, δεν ξέρω, όλοι οι εκπρόσωποι μας θα πρέπει να έχουν και αυτό το καθήκον. Και αυτή την ταινία θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην εξωτερική μας πολιτική. Εδώ στην Ευρώπη δημιουργήθηκε αυτό το μέσο που δείχνει την ευρωπαϊκή άποψη. Που δείχνει ότι έχουμε φιλοξενήσει στο ευρωπαϊκό έδαφος και ξένους πολιτισμούς. Και όλα αυτά πρέπει να τα προβάλλουμε, να τα προβάλλουμε και προς άλλες χώρες. Θα προσπαθήσω να κάνω μια πρόταση, δεν ξέρω αυτό το πετύχω, όχι για ένα Erasmus Plus μόνο, να έχουμε και ένα μέσο πολύ συγκεκριμένο που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε για την πρόταση του πολιτισμού. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε το λόγο. Λοιπόν, 5 Δεκεμβρίου... Α, όχι, μισό λεπτό. Η κυρία Μπίλτερ από την Επιτροπή. Σας ξέχασα, συγγνώμη. Θέλετε... Α, είστε από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θέλετε να πείτε κάτι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σας ξέχασα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είμαστε από αυτό ε, το οικοδόμημα, το αναποτελεσματικό άνευ που είπατε, αλλά τέλος πάντων χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε λίγο για το τι κάνουμε. Είχα προβλέψει να σας πω σε τρία σημεία πώς εμείς ε, συμμετέχουμε στην ε, διαπολιτισμική ανάπτυξη και πώς και εμείς η ΑΕΔ βρίσκουμε ε, το χώρο μας σε, σε, αυτόν τον κόσμο που η ταυτότητα, η θρησκεία, ο πολιτισμός έχουν μεγάλη σημασία και να σας πω ότι και εμείς ήρθαμε σε επαφή με ένα project ε, που βοηθά και αξιοποιεί προγράμματα ανταλλαγής όπως το Εράσμους τρία σημεία. Τέλος πάντων τα δύο θα τα δω πολύ σύντομα γιατί είναι περασμένη ώρα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει η μηδιάδα πρωτοβουλειών και εμείς προσπαθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. έχουμε κάποια μέσα στη διάθεσή μας και το Ίδρυμα Αναλίντ μεταξύ αυτών και προσπαθούμε από κοινού να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία αποφεύγοντας τις αλληλεπικαλύψεις. Επίσης είδαμε πως αυτά όλα οδήγησαν ε, ε, στη διασταύρωση αν θέλετε. Έχουμε τους επέφυνους μηχανισμούς μέσων για την ε, για το μετριασμό των διαφυλετικών εντάσεων και ούτω καθεξής. Έχουμε σε αυτό το τομέα και εισερχόμενους, έχουμε ένα κέντρο διαθρησκιακού διαλόγου στην Αυστρία, είχε ένα παγκόσμιο φόρουμ πρόσφατα, η εικόνα του άλλου λεγόταν, ε, ήταν ο τίτλος του. Και άλλες πρωτοβουλίες που μπορεί να μην εντάσσονται ακριβώς σε, αυτό το θέμα, αλλά για το πώς βλέπουμε ένα στον άλλο, ε, τα θρησκευτικά, η θρησκευτική παιδεία, πόσο σημασία έχει εντός και το σχολείο κτλ. κτλ. Ολοκληρώνοντας με το πρώτο λοιπόν θα έλεγα ότι εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τις να αυτό που μπορούμε να ενισχύσουμε τα θετικά. Δεύτερο, η θρησκεία είναι σημαντική και στην εξωτερική πολιτική. Αυτό δεν είναι καινούριο, αλλά ορισμένα κράτη-μέλη κατάλαβαν πια ότι η πολιτική βάση ταυτότητας αυξάνεται, όχι μόνο στην Ευρώπη και στον κόσμο, τον ευρύτερο. Εμείς παρακολουθούμε, επειδή στο γαλλικό σύστημα ήταν το πιο αστείο, έχει βάλει τα θρησκευτικά και το FCO και οι συνάδελφοί μας από την Ολλανδία μας βοηθάνε και αυτοί γιατί θέλουμε να εξοπλίσουμε του υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής για να αυξηθούν οι δεξιότητες ε, οι πολιτιστικές και στον τομέα της θρησκείας και όχι μόνο των γλωσσών. Και βλέπουμε και άλλους τομείς που αγνοούμε την θρησκεία. Κάποιες φορές ε, τη θρησκεία την περιορίζουμε στο θέμα της ε, ανεξιθρησκείας ή της ελευθερίας των θρησκευτικών πεπιθήσεων, που είναι ένα κομμάτι μόνο. Το ρόλο επίσης των θρησκευτικών φορέων ε, τον βλέπουμε πηγαίνοντας σε ε, χώρες που, και χώρους που δεν είχαμε επισκεφθεί μέχρι τώρα, πρόληψη συγκρούσεων, αντιπαθήσεων κτλ. Και όπως είπατε κι εσείς, θα πρέπει πραγματικά οι πολιτικές, οι εσωτερικές, εξωτερικές ε, να μην είναι απομονωμένες, αλλά να ε, επηρεάζουν μεν τις δε. Και ξέρουμε και ότι υπάρχουν και πολλοί φορεί ε, πολιτικοί που εμπνέονται από την ε, θρησκεία, όπω είναι και τα λοιπά υπάρχει το έργο του OIC. Θα σταματήσω εδώ με το δεύτερο σημείο, λέγοντα ότι έχει ρόλο η θρησκεία. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αρχίσαμε να οργανώνουμε και εκπαιδευτικά μαθήματα για το προσωπικό μας και για τα κράτη-μέλη. για να καταλάβουμε τις ε, σημαντικότερες θρησκείες, δίνουμε έμφαση ιδιαίτερη βέβαια στο Ισλάμ, σχέση πολιτικής και θρησκείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μελέτη του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας και θρησκείας, εκοσμίκευση και όταν κάποιο είναι αποσπασμένο στο εξωτερικό από το προσωπικό μας να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα. την επικοινωνία, ε, την άμεση, δεν την αντικαθιστά τίποτε. Μόνο έτσι μπορούν ε, να, σπάσουν τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις ε, και να υπάρξει καλύτερη γνώση. Η... Το Εράσμος ήταν μια επιτυχημένη ιστορία και είμαστε υπερήφανοι. Εκτός όμως από αυτή την ανταλλαγή έχουμε και κάποιους εδώ καλύπτει μόνο το 1% δυστυχώ Έχουμε και τις λεγόμενες εικονικέ ε, ανταλλαγές, virtual exchange. Μία μη κερδοσκοπική ομάδα από τι ΗΠΑ ξεκίνησε, είχε έρθει εδώ το Μάιο, είδε το Connect, είδε το Education and Culture, Του φέραμε να δουν το κοινοβούλιο, δεν ξέρω ποιο υποδέχθηκε, τέλο πάντων ήρθαν εδώ στο κοινοβούλιο και θέλω να σα πω ότι η ιδέα τους ήταν ότι αντί να έχουμε μια βαθιά ανταλλαγή μεν, αλλά με λίγους ανθρώπους, προνομιούχους, αυτοί άλλαξαν τα πράγματα, αντέστρεψαν αυτή τη στήλη αν θέλετε, ώστε μέσω διαλόγων εντός ενός εξαμήνου πάνω από 100 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν και τι έκαναν τελικά. μελέτησαν ε, τα επιπτώσεις αυτού του προγράμματος ανταλλαγών. Τι αντιλήψεις είχαν οι συμμετέχοντες πριν και μετά. Και είναι και πιο φθηνό αυτό το πρόγραμμα. Έχοντας πολύ ευρύτερο ε, στόχο. Φτάνει στις γυναίκες του κόλπου, στις γυναίκες Αιγύπτου. Ε, μπορείς να αυξήσεις ακόμη περισσότερο το ρόλο των προγραμμάτων ανταλλαγής όπως το Εράσμους. Εμείς παρακολουθήσαμε και από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης πάρα πολύ προσεκτικά αυτό το πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνέλευσης του ΟΗΕ. χρηματοδοτήθηκε από την οικογένεια του θανόντος πρέσβη Στίβεν ο Ευρωπαϊκών, που δημιούργησε ένα ταμείο, ένα ίδρυμα. Εμείς ε, δώσαμε την πολιτική μας ευλογία σε αυτό και μάλιστα με χορηγία 5 εκατομμυρίων. Και θέλουμε να δούμε πώς εμείς μπορούμε ως Ευρωπαίοι και τους φοιτητές μας να τους διασυνδέσουμε, αλλά να βάλουμε στη, στα κεφάλια μας και στο θεματολόγιο μας και αυτή την έννοια της εικονικής ανταλλαγής για μεγαλύτερη γνώση μεγαλύτερες διαπροσωπικές ε, πολιτισμικές δεξιότητες, ε, να ε, ξεχάσουμε τις εύκολες λύσεις και τη, τη ριζοσπαστικοποίηση της νέας γενιάς. Βέβαια δεν αντικαθιστά η άμεση, δεν μάλλον υποκαθίσταται η προσωπική άμεση επαφή και γνώση, αλλά Τέλο πάντων, έχω να σα δώσω και περισσότερε πληροφορίε για αυτό το πρόγραμμα, αν σα ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, καλό είναι που δεν σας ξέχασα τελείως. Ε, ήρθατε εδώ καλά προετοιμασμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καλό είναι που η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, ε, παρευρέθηκε και μας είπε αυτά που είχε και τα είχε προετοιμάσει και τόσο καλά. Αν θέλετε στείλτε μας υλικό για το πρόγραμμα ανταλλαγής για το οποίο μιλάτε και με χαρά μας θα το προωθήσουμε και θα το διαδώσουμε. Ε, δεν έχουμε μόνο το πρόγραμμα Erasmus+, Plus, έχουμε πολλά επίπεδα. Ε, για τους νέους έχουμε ένα ειδικότερο πρόγραμμα και για την λαϊκή επιμόρφωση έχουμε προγράμματα αδελφοποίησης. Είναι παρόμοια και είναι κάτι που το κάνουμε με χώρες ε, σε όλο τον κόσμο. Και είναι σημαντικό το ότι έχετε και ένα ταμείο από το οποίο μπορείτε να βρείτε χρηματοδότηση. Πραγματικά αυτές οι ανταλλαγές βελτιώνουν και ενισχύουν την αίσθηση ότι ζούμε με άλλους πολιτισμούς, συμβιώνουμε και με άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ίσως μπορούμε να σας στείλουμε και κάποιες ιδέες ε, στην Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ίσως μπορούμε να υποβάλουμε και κάποια τροπολογία με αυτό στο νου. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό στις 5 Δεκεμβρίου. Ε, είναι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Και θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τη στρατηγική έκθεση 2013 για την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής είναι η αρμόδια επιτροπή. Bitte, Με συγχωρείτε, η Επιτροπή Αναφορών είναι η αρμόδια επιτροπή. Νομίζω ότι δεν αποτελεί μυστικό το ότι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις ε, ε, όσον αφορά την ε, δημόσια στήριξη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι από εσά θα συμφωνήσετε ότι υπάρχουν πολλές παροχές και η έκθεση 2013 για την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σίγουρα αναδεικνύει το, προνόμιο του να είναι κανείς Ευρωπαίος πολίτης. Ε, εξακολουθούμε όμως να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις. Ε, οι περισσότεροι πολίτες όμως δεν έχουν ιδέα τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Ε, στις περισσότερες περιπτώσεις γνωρίζουν μόνο τα βάρη που τους επιρρύπτονται και που προέρχονται από τις Βρυξέλλες θα πρέπει και υπάρχει αυτή η διαδεδομένη προκατάληψη ε, και σίγουρα το βλέπω και εγώ στη Δανία, στη δική μου εκλογική περιφέρεια ότι όποτε υπάρχει ένα πρόβλημα το φταίξιμο πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ασφαλώς η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά για να βοηθήσει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους και προσπάθησα να το δω το θέμα αυτό στην έκθεσή μου. Να τονίσω, να αναδείξω δύο, σημαντικά, δύο σημαντικούς τομείς. Ε, την επίγνωση, την ευαισθητοποίηση, παράγραφος 1 ε, ήδη υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες, επιτάπητος. Ασφαλώς όμως δεν αρκούν αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής. Πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας και να ε, μας βοηθήσουν και τα κράτη-μέλη. Ε, αυτό μπορούμε να το φέρουμε με τροπολογίες ε, τη στιγμή που έχουμε τόσες πολλές ε, σειρές. Η παράγραφος 4 έχει να κάνει με τη σημασία της υποστήριξης των πανευρωπαϊκών δικτύων, το δεύτερο στοιχείο. Θα θυμάστε ότι είχαμε κάποια προβλήματα όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξαφνικά ακύρωσε την προκήρυξη διαγωνισμού στο διαδίκτυο. Το έκανε αυτό χωρίς να μας συμβουλευτεί. Ε, πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω στο θέμα αυτό. Αυτά θα πω, Πρόεδρε. Ε, ανυπομονώ να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και να ανταλλάξουμε άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι με μεγάλη μου χαρά μιλάω σήμερα για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, γιατί και εγώ συμμετείχα στην Επιτροπή Αναφορών ως σκιώδης εισηγητής. Υπάρχουν κάποια θέματα που ξέρουμε για την ηθαγένεια των πολιτών και υπάρχουν και κάποια νομικά ζητήματα που πρέπει να δει η Επιτροπή Αναφορών. Όμως, για να ε, παραθέσω και αυτά που είπε ο συνάδελφος. Ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό το να ενθαρρύνουμε την ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα εδώ και αυτό θέλουμε να προωθήσουμε. Και να σας πω και τη δική μου προσωπική άποψη που πάει λίγο παραπέρα. Είναι μια, έχουμε μια καλή ευκαιρία εδώ να προσεγγίσουμε ε, αυτό το θέμα ως ε, πολιτικό, ή να μιλήσουμε για την πολιτική εκπαίδευση των Ευρωπαίων πολιτών. Και νομίζω ότι είναι καλό να δούμε εδώ και την ε, εκπαίδευση και κατάρτιση και των καθηγητών. να μην ξεχάσουμε τη σημασία αυτού του θέματος εδώ. Έχουμε ε, φέρουν μεγάλη ευθύνη εδώ τα κράτη-μέλη και ίσως ε, μερικές φορές προσπαθούν να αποφύγουν αυτή την ευθύνη, δεν καταβάλουν αρκετές προσπάθειες ε, για να βοηθήσουν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικασίες, να καλύψουν τέτοια ζητήματα. Όπως και να είναι, εγώ Χαίρομαι που έχουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και, το στηρίζω το σχέδιο. Ευχαριστώ, Σαντιάγου. Ε, Ευχαριστώ, Ντόρι. Ευχαριστώ και τον Μόρτεν την γνωμοδότηση. Θα ήθελα να επιμείνω στα εκλογικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ε, που διαμένουν σε τρίτη χώρα όπως στην Ισπανία. Και έχουν δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές εκλογές, χωρίς να είναι όμως εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Και πολλοί ενδεχομένως δεν γνωρίζουν αυτό τους το δικαίωμα. Θα ζητούσα λοιπόν να δούμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα, αφού έχουμε σύντομα τις ευρωεκλογέ να, γίνει, να γίνει, να διοργανώσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση, ώστε αυτά τα άτομα να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να μπορέσουν να ασκήσουν ε, το δικαίωμα ψήφου στην τρίτη χώρα στην οποία διαμένουν, γιατί πολλές φορές δεν το γνωρίζουν, μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι και να μην γνωρίζουν ακριβώς ε, τι πρέπει να κάνουν. Ή μπορεί να είναι άτομα που δεν έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση ή επαφή με το διαδίκτυο. Θέλουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή σε ευρωεκλογέ. Λέμε ότι είναι, είναι μικρή προσέλευση ευρωεκλογέ και μα ε, ενδιαφέρει αυτό. Γιατί να μην κάνουμε κάτι λοιπόν και προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θα έλεγα ότι σήμερα έχουμε μια Ευρώπη που είναι δημοκρατική και διαφανής, είναι μια νέα Ευρώπη που είναι κοντά στους ε, πολίτες της και αυτό είναι κάτι θετικό. Ο Σαντιάκο μίλησε για τα δικαιώματα ψήφου, ε, για, την, για τα δικαιώματα οικουμενικής ε, ψηφοφορίας. Έχουμε πολιτικά δικαιώματα, κοινωνικά, οικονομικά δικαιώματα τα οποία εγγυόμαστε. Είναι θεμελιώδη δικαιώματα αυτά που αφορούν ελευθερίες και παρατηρούμε σήμερα ότι υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στην Ευρώπη και στους πολίτες και ότι η γνώση δεν αυξάνεται, υπάρχουν κάποια πολιτικά κινήματα που ε, είναι προς το συμφέρον τους να παραμείνουν έτσι τα πράγματα. Ο Μπέκερ μίλησε ε, για, τα, για τις αιτήσει που μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες, για τις αναφορές. Και συνειδητοποιούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και ιδιαίτερα ε, στους προσεχείς μήνες πρέπει να τους ευαισθητοποιήσουμε ε, ως προς το τι θετικό μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη. Όπως ξέρετε η εικόνα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ καλή και όλοι θεωρούν ότι όλα είναι από πρόβλημα που προκύπτει από την Ευρώπη. Ε, και εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω και για κάποια εθνικά σχέδια μέσα στα κράτη-μέλη, γιατί, γιατί έτσι είμαστε πιο κοντά στους πολίτες. Γιατί μερικές φορές ε, σε εθνικό επίπεδο τα κράτη-μέλη όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά ρίχνουν το φταίξιμο στις ευρωπαϊκές αρχές Επομένως, ε, χαιρετίζω ιδιαίτερα τις ε, αναφορές που έγιναν για εκπαίδευση των ε, καθηγητών, για ευαισθητοποίησή τους ως προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί αυτοί είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν μια πιο θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα παιδιά, στους νέους. Και αυτό θα αυξήσει την την εικόνα, μια καλύτερη εικόνα της Ευρώπης. Κύριος Ρέπο, ευχαριστώ. Α, το κείμενο αυτό είναι πάρα πολύ καλό. λέμε πώς μπορούν να προστατευθούν καλύτερα και να αντικατοστούν καλύτερα τα δικαιώματα των πολιτών. Μιλάμε για το Europe Direct και το Your Europe. Ε, το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα εργαλεία δεν είναι αρκετά γνωστά. Οι περισσότεροι πολίτες δεν γνωρίζουν ε, αυτά τα μέσα που είναι στη διάθεσή τους και επομένως δεν τα χρησιμοποιούν. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να ασχοληθούμε με την ευαισθητοποίηση ε, ε, των πολιτών προς τα μέσα που είναι στη διάθεσή τους. Ε, ένα δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι για το πρόγραμμα, για τα ευρωπαϊκά πρόγραμματα για τους πολίτες. δώσαμε μια έγκριση στην τελευταία ολομέλεια και ο στόχος είναι εδώ να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τις αξίες της Ευρώπης, ε, τον πολιτισμό και την ιστορία. Θέλουμε να ανοίξουμε μια συζήτηση, να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Έτσι θα φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και θα τους δώσουμε ένα κίνητρο για να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Πρέπει να αλλάξουμε τις νοοτροπίες. Και δεν μιλάω μόνο για τους πολιτικούς εδώ, μιλάω για όλο τον κόσμο. πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες πώς διεξάγονται οι στρατηγικές σε εθνικό ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, βλέπετε και από το έγγραφο αυτό ότι στο πολίτες ε, δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπετε θα μειωθεί πάλι η χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα νητικό, ένα δύνατο σημείο Χρειαζόμαστε όμως τους πολίτες, τους χρειαζόμαστε και πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι χρειάζεται η εμπλοκή τους, ε, είναι η δική τους Ευρώπη. Και ταυτόχρονα θα μειωθεί ο προπολογισμό ε, ε, για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες κατά 12% ο νέος προϋπολογισμός θα έχει μόνο 160 εκατομμύρια για 7 χρόνια και για 27 κράτη-μέλη. Δηλαδή λιγότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ ανά και ανά Ε, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. εμείς πιστεύουμε στην, στο μέλλον της Ευρώπης, ε, Πρόεδρε, και πρέπει να το δείξουμε αυτό και στους πολίτες. Ναι, ε, έχετε δίκιο και πρέπει να είμαστε ε, έτσι ενθουσιώδεις, αλλά μη θυμώνετε με εμά, δεν τα έχουμε αποφασίσει εμείς αυτά. 5% θα είναι η μείωση και υπάρχουν και αρκετοί αρχηγοί κρατών που δεν συμφωνούν με αυτές τις περικοπές κάθε φορά λέμε ότι πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια όρια. Απλά πρέπει να, περάσουμε, γυρίσουμε στις χώρες μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ε, βέβαια, αυτό δεν είναι αρκετό. δεν χρειαζόμαστε πολλά κονδύλια και δεν ξέρουμε από πού μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά τα λεφτά. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όμως μόνοι μας, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ως ομάδα για να ε, φέρουμε μια αλλαγή στην Ευρώπη. Ναι, έχετε ε, δίκιο, πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το σωστό. Αλλά δεν μπορεί ο Επίτροπος να πείσει τους ε, ψηφοφόρους ε, στην, στην κάθε εκλογική περιφέρεια. Αυτό θα το κάνετε εσείς και εγώ. Πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καθένας ε, τους πόρους που έχει στη διάθεσή του για να περάσει αυτό το ευρωπαϊκό μήνυμα και πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν χρήματα και για αυτό το πράγμα. Αυτό όμως θα το αποφασίζουν οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων. Και, και τώρα, κύριε Μπέκερ, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να ζητάτε κάτι που ήδη υπάρχει. Έχουμε ήδη το Erasmus Plus. Όχι το, το Erasmus, το Erasmus Plus. Ήδη έχουμε εκεί κάτι για την εκπαίδευση, ε, για ανταλλαγή καθηγητών ε, και γενικά για όλων όσων δουλεύουν στην, στον τομέα της εκπαίδευσης. Ε, το ξέρετε, το έχουμε ήδη αυτό και πρέπει να το γνωρίσουν όλοι δεν σας κρύβω και το γεγονό ότι και εγώ ήμουν καθηγήτρια και εσείς ε, νομίζω και ο κύριος Λόκενγκάρν. Ναι, ε, πρόεδρε, πήρατε τα λόγια από το στόμα μου. Και εγώ θα ήθελα να πω στον κύριο Μπέκερ ότι ότι αυτά είναι θέματα που ήδη έχουμε συζητήσει για το Erasmus Plus όπως και να έχει πάντως, ε, σας ευχαριστώ που υπογραμμίσατε αυτό το σημείο για το ρόλο των καθηγητών. Ε, όντως παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και ευτυχώ έχουμε αυτό το πρόγραμμα Erasmus Plus και καταφέραμε μέσα στις διαπραγματεύσεις να κάνουμε κάτι για τους καθηγητές. Ε, έχουμε λοιπόν κάτι, αλλά σίγουρα μένει ακόμα δουλειά και άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν. κύριε Φίσας, για τα δικαιώματα ψήφου, όντω μπορούμε να έχουμε μια τροπολογία εδώ να... που θα ασχολείται με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό με αυτό που θίξατε. Ιδιαίτερα βλέποντας ότι έχουμε ενόψει, ε, ενόψει μας τις και ε, ήδη το Κοινοβούλιο έχει μια πολύ φιλόδοξη ε, εκστρατεία και νομίζω ότι όλοι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν ξέρω πού θα φτάσουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ε, ότι αυτό το ε, θέμα αξίζει. Στην Δανία είχαμε τοπικές εκλογές και ήταν πολύ δύσκολο να ε, πείσουμε τους νέους να συμμετάσχουν. Είχαμε πολύ καλές εκστρατείες στη Δανία και τελικά τα θυμητικά στοιχεία ήταν καλύτερα είχαμε μία αύξηση της τάξης του 5 με 7% ε, χάρη σε αυτή την εκστρατεία που κάναμε. Άξιζε λοιπόν ε, τον κόπο και νομίζω ότι πρέπει να μιμηθούμε αυτό το καλό παράδειγμα ε, και να δείξουμε ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε τέτοιου είδους εκστρατείες και τέτοιου είδους προσπάθειες. Επίσης, συμμερίζομαι αυτήν την άποψη του κύριου Ρέπο. Πρέπει να αλλάξουν όντως οι νοοτροπίες. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε πολλές καλές πρωτοβουλίες και έχουμε και ε, μία για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και για αυτά που οι άνθρωποι συνήθως βρίσκουν βαρετά, αλλά για, τα, για όλες τις υπόλοιπες πτυχές και νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε αν θέλουμε να αυξήσουμε την ε, ε, ενημέρωση, αν θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και να τους μιλήσουμε ως ε, Ευρωπαίοι. Εκεί μπορούμε να βασιστούμε να εμπλουτίσουμε το λόγο μας και να πούμε τι μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι για τον κόσμο. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία εδώ και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, έχουμε πολλές καλές οργανώσεις και εκδηλώσεις ε, παντού στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας και τις συνεισφορές σας και αν να δω τις τροπολογίες που θα υποβάλλετε. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης θα βοηθήσει με την πίεση που θέλουμε να ασκήσουμε. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και νομίζω ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες ε, ουσιαστικές σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μπορείτε για τις τροπολογίες, ή μάλλον πρέπει να τις στείλετε μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο 11 δεν ξέρω, δεν, αν έχετε καμία αντίρρηση με την απόφαση των συντονιστών. Αν δεν τις ξέρετε, δεν πειράζει. 12 διάφορα, δεν υπάρχουν ε, διάφορα. Ε, ή μάλλον εγώ έχω κάτι να πω για το βραβείο Λουξ. Να το δείτε και να α, ψηφίσετε. Ε, ε και, και να μιλήσετε και στους συναδέλφους σας, όλοι σας όλοι σας να το ζητήσετε από τουλάχιστον άλλους πέντε συναδέλφους. Η, η πρόεδρος ευχαριστεί και τους ε, διερμηνείς και εμείς σας ευχαριστούμε και επόμενη συνεδρία στη 17 Δεκεμβρίου.